Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία, να σα ρωτήσω αν έχετε αντιρρήσει και να εγκρίνουμε κατευθείαν την μερίσια διάταξη όπω σα έχει μοιραστεί. Υπάρχουν αντιρρήσει, Όχι. Θεωρούμε ότι εγκρίθηκε. Και σα προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ε, περασμένης ενάτης τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης 9 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία λοιπόν. Θεωρούμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά τη προηγούμενη συνεδρίασης. Και σα θυμίζω ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Ως ήθιστε. Θα περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στην ψηφοφορία τη έκθεση. την τελική τη μορφή. Ε, ο εισηγητή μα, ο κ. Γιακολίνο, επέβαλε το σχέδιο εκθεσή του στην ε, περασμένη συνεδρία στις 18 Ιουνίου και έπειτα από τους συναδέλφους υποβλήθηκαν 392 τροπολογίες. Ο εισηγητής και οι σκιώδης αλλά και οι συντονιστές και όλοι οι συνάδελφοι που προσπέγραψαν αυτές τις τροπολογίες συμμετείχαν σε ομαδικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να μελετήσουν και να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε συμβαστικές λύσεις. Και η Γραμματεία συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια και όλο αυτό το έργο οδήγησε σε 24 συμβαστικές λύσεις που θα πρέπει να ψηφιστούν μαζί με την τελική μορφή της έκθεσης. Εδώ έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γιακολίνο, θα του δώσω αμέσως το λόγο επειδή είναι ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς μερικές διευκρινήσεις. Συγκεκριμένα στον κατάλογο των ψηφοφοριών, η τροπολογία 127 και 195 δεν θα έχουν πλέον μείον δίπλα τους. 127 και 195 με συν έπειτα στη συμβιβαστική 2 μετά την ανακύκλωση χρημάτων να προσθέσουμε βάση των αρχών της αλληλεγγύης και επικουρικότητας. Και στη συμβαστική λύση, στη συμβαστική πρόταση 6, εκεί που αναφέρεται η αρχή της αναλογικότητας, λείπει και της επικουρικότητας. Προστίθεται το και της επικουρικότητας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Γιακολίνο. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι, όχι αλληλεγγύη, επικουρικότητα και αναλογικότητα. Δεν είναι η στιγμή σε αυτή την ε, συνεδρίαση να μιλήσουμε για αλληλεγγύη. Δεν χρειάζονταν η διευκρίνηση. Αλληλεγγύη θα είμαστε και ούτω ή άλλω ε, η δική σα δουλειά είναι μέγιστη σημασία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να σα θυμίσω να κοιτάξετε αν έχετε τι κάρτε ψηφοφορία σα. Τι έχετε. Ωραία. Ψηφίζουμε την ε, συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έπειτα, τροπολογία 98, 98. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. αυτό έχουμε. Ψηφίζουμε την 99. 99. Ψηφίσατε άπαντες. Όχι, να διορθώσω. Δύο λεπτά.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 Σε ξεχωριστή ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε τώρα τη συμβαστική συνολικά και μετά θα δούμε τις διάφορες κατατμήματα ψηφοφορίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Τώρα, προτεραιότητας. Προτεραιότητα 7. Πέρας. Δεν ψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. Προτεραιότητα 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προτεραιότητα 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προτεραιότητα 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προτεραιότητα 14. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελευταία προτεραιότητα, η 15η. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 104 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 107 έχει αποσυρθεί. 105 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. <coughs> Απορρίπτεται. 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 τώρα, συμμεβαστική 23. Τρε, τρεις ε, ξεχωριστές ψηφοφορίες. Ξεκινούμε με την πρώτη. Ξεχωριστή από την αρχή της τροπολογίας ως το Law Agency εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, από το fraud μέχρι το calls on the commission και unaccompanied minors. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εψήφισαν παντέ Εγκρίνεται. Τελευταία ξεχωριστή ψηφοφορία αυτής της συμβαστικής λύσης. Calls on the Commission έως, έως το τέλος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκατόν τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 369. Άρχεται. 369. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 127. Μετά θα ψηφίσουμε την 128 μας. Η γραμματεία μου επισημαίνει ότι πρόκειται για δύο συμβατές τροπολογίες. 127, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 128, άρχεται η ψηφοφορία. 128. Πέρας. Εγκρίνεται. 129. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Από την αρχή ως το trade unions. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη ξεχωριστή ψηφοφορία, υπόλοιπη τροπολογία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίτεται. 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 204, 204 τώρα, τροπολογία 204, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 138, 138, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Οπότε πηγαίνουμε στην 141. 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 142. 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 144. 144. Άρχεται η ψηφοφορια Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 145-145. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ένα λεπτάκι κυρία Μακοβέη. noi procediamo con il voto, andiamo all'emendamento... Προχωρούμε με την τροπολογία 1 5 135, όχι, 1 Όχι 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 147-147 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 149 και 147. Δύο τροπολογίες πανομοιότυπες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν λειτουργεί. Ξαναψηφίζουμε την 149 και 187. Πανομοιότητες οι τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκατόν ογδόντα οκτώ. Ένα Άρχεται η ψηφοφορία. Εκατόν ενενήντα. Εκατόν πενήντα, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 152-152. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 133. 133. Πέρας. μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. 29 μάλλον θα είναι η πλειοψηφία οι αρνητικέ ψήφοι. Απορρίφθηκε. Μάλλον. 154 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 155. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 156. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 157. 158 Εκατόν 158-158, 158, με ξεχωριστή ψηφοφορία. Μέχρι το, το, το, η πρώτη ψηφοφορία είναι από την αρχή μέχρι το Mafia Type Assets. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα από το Σάτσα στο τέλος. Πέρας. Εγκρίνεται. 160... 159. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 160 161. 160. 160. Πέρας. Αγκρίνεται. 161. 161. η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 162. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 163 τώρα. 163. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. 154. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συμβαστική 7 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 167. 167. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 168. 168. Πέρας. Απορρίφθηκε. 169. Ε, αποσύρθηκε. 170. Άρχεται ψηφοφορία. 171 τωρα 1-7-1 τώρα. 171. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Τάνια εντάξει. Πέρας. Απορρίφθηκε. 1.35. 135 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 175 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 182. 182. 182 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα 183. 183. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 184. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 1.85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 189. 1.89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 191-9-0. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 191. 191. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 193, γιατί το 192 είναι πανομοιότυπο με, το, είναι πανομοιότυπο με την 191. 193 κατά τμήματα ψηφορίας, πρώτο τμήμα από την αρχή ως το At least Nationally. Ψηφίζουμε πρώτα αυτό το κομμάτι, ε, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Από το In Addition ως το τέλος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 194. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 195. 195. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 196. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 197. Άρχεται η ψηφοφορια Πέρα Πέρας. Απορρίφθηκε. 198-198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Αγκρίνεται. Τώρα, 200. 2-0-0. Il voto è chiuso. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 201, 201. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 202, 202. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 203. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 205. 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 206. 206. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 208. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική 9 μάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 210. 2-1-0. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 213, 213. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 214. 214. Άρχεται η ψηφοφορία. περα Απορρίπτεται. 215. 215. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 216. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 217-217. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία 218. 218. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ...219. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 220. 220. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 221. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 222. 222. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 223. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ...223. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφο... 226. 226. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 227. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσαμε. Απορρίφθηκε. Η 228. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Πάμε τώρα στην 229. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική 11. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην 2.34. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε. 2.35 ε, σε τμήματα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα που λέει including in cases, Φίνο ε, is inadequate. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 2.36. Και εδώ ψηφίζουμε σε τμήματα. Από εκεί που λέει recommends a μέχρι criminal activities. Ψηφίζουμε για το πρώτο κομμάτι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε αυτό το πρώτο κομμάτι και ψηφίζουμε τώρα για το δεύτερο, including by, μέχρι Common Action Plan. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την 12. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πάμε στην 374. Στην 374. Λοιπόν, 374. Ε, ψηφίζουμε σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Από εκεί που λέει expresses concern μέχρι for criminal organizations. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση στα γαλλικά. Εντάξει, ακούτε γαλλικά. Έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Από εκεί που λέει have a particularly negative μέχρι those mentioned above. Ψηφίζουμε παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα. Έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην 238. Εδώ ψηφίζουμε μόνο για το δεύτερο τμήμα, γιατί το πρώτο τμήμα έχει καταπέσει. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα και όχι για το πρώτο. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για την 239. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 2.41 τώρα. Ψηφίζουμε για την 2.41. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την 242. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 2.46 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφορία. Τώρα, οι 2.47, 48 και 49 ψηφίζουμε ε, και για τις τρεις. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έκλεισε. Απορρίπτονται. Τώρα, για την 2.50 ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφορία. Ψηφίζουμε για την 2.51 παρακαλώ. για την 252. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 254. Έκλεισε η ψηφορία. Ψηφίζουμε για την 254. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική 14. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και περνάμε τώρα στην 258. Ψηφίζουμε για την 258. Έκλεισε. Ψηφίζουμε για την 259. Ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε. Η 260 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε για την 261. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την 262 παρακαλώ. τμήματα 2.63 σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι όλο το κείμενο χωρίς το financial and criminal. Ψηφίζουμε για αυτό το πρώτο κομμάτι. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το δεύτερο τμήμα, εκεί που λέει Financial and Criminal, ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 264. Πάμε στην 265. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 268. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 269. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 270. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Τώρα πάμε στην 275. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.76. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.77. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε για μία που μας ξέφυγε, η 271. Ψηφίζουμε για την 271. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 2.72. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 273. Ψηφίζουμε. Για την 273 έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, για την 274 ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε για την 278. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 279. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 280. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 281. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 281. Μπερδεύτηκε η πρόεδρος. 282 νους. Ψηφίζουμε για την 282. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 283. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Πάμε στην 286. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 287. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 288. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 289. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην συμβαστική 15. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 294. Παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Λοιπόν, πρέπει όμως ε, να ξαναψηφίσουμε για την 294. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 296. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.97. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 2.98. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την 299. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα για την 300. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Τρία μηδέν τρία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πάμε τώρα στην 304. 304. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 305. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα για την 306. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 307 και 308. Ε, είναι ίδιες ακριβώς τροπολογίες. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 310. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 311. Ε, Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία εγκρίνεται. Στην 312 ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 313. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 314. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την συμβαστική 16. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 3.20. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 321. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. επαναλαμβάνουμε την τροπολογία, αλλά η γραμματεία ε, πολύ σωστά μου λέει να αφήνω λιγάκι χρόνο να ψηφίζετε. Κατόπιν τούτου ψηφίζουμε για την 321. Η 320 απορρίφθηκε. Έκλεισε η ψηφοφορία για την 321. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα για την 322. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε για την 323. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 326. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 326. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κατόπιν οι επόμενες δύο, οι 27 και 28 μοιάζουν, γι' αυτό ψηφίζουμε ε, από κοινού για την 327 και την 328. Ψηφίσατε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την 329. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 330. Ψηφίζουμε Έκλεισε η ψηφορία. Τρία Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την 332. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 3.33 τώρα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 3.34. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική 17. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 3.40 τώρα. Ψηφίζουμε για την 3.40. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 341. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 342. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και βλέπω ότι από το ΕΛΚ ε, χαμογελούν. Τώρα ψηφίζουμε για την 343. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 344. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 345. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για δύο ακριβώ ίδιε τροπολογίε, την 346 και την 347. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 351. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 352 απορρίφθηκε. 353. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα, 3.54. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται για την 3.55 τώρα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 356. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 357. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Για την 367. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται και τώρα ε, για την 368 ψηφίζουμε σε δύο τμήματα εκεί που λέει ε, calls on the commission will ε, wildlife trafficking ψηφίζουμε παρακαλώ για αυτό το πρώτο κομμάτι έκλειση ψηφοφορία εγκρίνεται και για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε τώρα για το δεύτερο τμήμα, ε, εκεί που λέει Highlighting Clear Plants and Trees into the Union. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα αυτής της τροπολογίας. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην 3.75. Ε, Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 385. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 386 ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 388. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, ψηφίζουμε για την 389. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα, έχουμε μία προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω αν έχετε αντιρρήσεις. Αν όχι, μπορούμε να ψηφίσουμε για την προφορική τροπολογία με βάση το κείμενο που έχετε μπροστά σας. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πρέπει να ε, επαναλάβουμε την ψηφοφορία γιατί ένα συνάδελφος από το ΕΛΚ περισσεύει. Σε αυτή την αίθουσα είναι πάρα πολύ οι συνάδελφοι του ΕΛΚ. Παναλαμβάνουμε λοιπόν ε, αυτήν την προφορική τροπολογία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε στην 390. Ε, Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 391 αποσύρθηκε. 392 τώρα παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και ξεκινάμε με τα εκτιμώντας. Η τροπολογία 1 παρακαλώ. έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Οι δύο, εκτιμώντας δύο. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τρία αποσύρθηκε. Η τέσσερα ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πέντε. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία εγκρίνεται. Η 6. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 7. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προφορική. Μάλλον ε, τροπολογία 8. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Και άλλη μια προφορική τροπολογία, δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίρρηση, όχι από ό,τι βλέπω, άρα ψηφίζουμε επί του κειμένου, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται, προφορική τροπολογία υπαριθμών 3, διαφωνεί κανείς, όχι, προχωράμε λοιπόν, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ή για την 4 την προφορική έχετε αντιρρήσεις. Όχι, ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Ε, από ό,τι βλέπω δεν έχετε αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε. Ε, η ψηφοφορία είναι ανοιχτή. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 9. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 10. Ψηφίζουμε. είναι η τέταρτη φορά που επαναλαμβάνουμε μια ψηφορία. Κοιτάξτε, εγώ δεν βιάζομαι. Ε, το ξέρω ότι κουράζουν οι ψηφορίες, αλλά αν έχετε καλοσύνη να προσέχετε λιγάκι. Σας παρακαλώ. Πού ήμασταν τώρα. Η τροπολογία η 10. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε πρώτα την 9. 9. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Λάθος, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 11. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται. Η 12 και η 13 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε και για τις δύο. Ψηφίζουμε για τη 12 και τη 13. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Περνάμε στην συμβαστική 18. Ξέχασα τη 14, λέει. Ψηφίζουμε για τη 14. Έκλεισε η ψηφορία. Απορρίφθηκε. Πάμε στην συμβαστική 18. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 19. Ψηφίζουμε για τη 19 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται 20. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Ψηφίζουμε για την συμβιβαστική 19. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία υπαριθμών 24. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 25 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 26. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε για την 27. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 28. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 29. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Il Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 3-4. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Να απορρίπτεται. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 37. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. περα Εγκρίνεται. Δύο τροπολογίες τώρα, πανομοιότυπες. Όχι, με συγχωρείτε, 38 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο πανομοιότυπες τροπολογίες, 39 και 40. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτές τις δύο τροπολογίες. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4-1, 41. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. 4-4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 46. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αποσύρθηκε 61, 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 20, συμβιβαστική 20, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 67, 6-7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 69. 6-9. έρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 70, 70-70 πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Πέρας. 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εβδομήντα έξι. Ε, επτά έξι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα δύο πανομοιότυπες τροπολογίες. τις ψηφίζουμε από κοινού, 78 και 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα γλωσσική αλλαγή. Όχι. Όχι. Περνάμε στην 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 81. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. 85, 85, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 87. 86 με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τοπολογία 86. Πέρας. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 τώρα, 8-9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ενενήντα τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 92 τώρα. 9-2. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. 9-3. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. αντιρρήσει. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο της προφορικής τροπολογίας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 95 κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα από το We the Judicial Independence ως το Interest. Ψηφίζουμε αυτό το πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεύτερη. Κατά τμήμα ψηφοφορία. Where is life discretion. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Allora adesso... Πολύ ωραία λέει η πρόεδρος. Ε, τώρα λοιπόν ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου όπως ε, τροποποιήθηκε το κείμενο. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 29 υπέρ, 0 κατά και 8 αποχές. δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή κύριο Γιακολίνο. Ε, μισό λεπτό γιατί ο κύριος Ταμπάρες θέλει να κάνει ε, επεξήγηση ψήφου. Κύριε Γιακολίνο, πρώτα θα προηγηθεί αυτή η επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, θα κάνω δηλώση ως ε, αντιπρόεδρος, αλλά για τους ε, σκιώδεις, για την ομάδα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, αλλά να πω ότι η ομάδα μας δεν μπορεί να ψηφίσει υπέρ, λόγω συγκεκριμένα μιας τροπολογίας την οποία κατέθεσε ο κύριος Κέρκοπ ε, για το PNR. Θεωρήσαμε ότι αν εγκριθεί ουσιαστικά θα έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συγκεκριμένα. Ε, το 52-3 λοιπόν ε, του εν λόγω κανόνα του Κοινοβουλίου η πράσινη ε, καταθέτουν ε, μία γνωμοδότηση μειοψηφίας η οποία θα πρέπει να επισυναυθεί στην ετολική έκθεση, ως ετολική έκθεση ουσιαστικά, στην έκθεση της Επιτροπής μας. Θα καταθέσουμε και τροπολογίες, αλλά ουσιαστικά αυτό που μας ενοχλεί είναι η τροπολογία Κέρκοπ. Συγκεκριμένα αυτή η τροπολογία μας ενοχλεί, άρα θα απόσχουμε τελικά. Έτσι λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να πω το εξή ότι επειδή σήμερα εγκρίναμε αυτό το ψήφισμα, κατ' ουσίαν σιγά σιγά τελειώνουν οι εργασίες αυτής της Επιτροπής της Ad Και στην Ολομέλεια, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου, θα ψηφίσουμε το τελικό ψήφισμα για τις εργασίες της ΚΡΙΜ. Είμαι λοιπόν στην ευτυχή χαρά να σας πω ότι το Προεδρείο ε, επέτρεψε να δημοσιευτούν αυτά τα έγγραφα, οι εργασίες οι οποίες καταλήξαμε στη διάρκεια των εργασιών μας μαζί με CD. Ε, ε, βέβαια αυτά όλα θα είναι στα αγγλικά, αλλά ε, θα μεταφραστούν ε, αργότερα και σε κάποιες άλλες γλώσσες. Αυτό το ε, πόνημα θα σταλεί σε όσους ενδιαφέρονται. Θα υπάρχει και ένας τόμος που όπως σας είπα αφορά τους τελευταίους 18 μήνες των εργασιών μας. Αυτό το έχει ήδη προετοιμάσει η Γραμματεία και μπορεί να σας το διανύμει σήμερα. Και τώρα ε, έχω την τιμή να δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή και κατόπιν στους αντιπροέδρους, ε, στους και όλους εισηγητές, σε όποιον τον ζητήσει. Συγχαρητήρια κύριε Γιακολίνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που κατέτσαν δυνατό αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα που αφορά την αντιμετώπιση της ε, μαφίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε, να αντιμετωπίσουμε, έχουμε μπροστά μας ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε και την δυνατότητα πλέον να ε, παρουσιάσουμε μία απάντηση στην ευρωπαϊκή πρόκληση Πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος ε, για την δουλειά που έχουν κάνει οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, ευχαριστώ την Πρόεδρο, τη ε, Γραμματεία, όλους εκείνους που θέλησαν να επισημάνουν τη σημασία όλης αυτής της υπόθεσης. Το θέμα της μαφίας είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Το ε, έγκλημα είναι κυρίως οικονομικό και τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν και οι συστάσεις ακολουθούν την ευταία κατεύθυνση. Ε, κληθήκαμε να καταρτήσουμε έναν κατάλογο συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και με βάση αυτές τις προτεραιότητες θα κρίνουμε συνεχώς ε, και την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και τις συγκεκριμένες δράσεις ε, στις οποίες θα προβαίνουν οι Επιτροπές αλλά και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Σε όλα τα κράτη-μέλη το θέμα του ε, μέλους της ε, μαφίας ε, πρέπει να προσδιοριστεί και αυτό έχει άμεση σχέση τόσο με το τραπεζικό απόλυτο όσο και με τις, ε, ε, τους τραπεζικούς παραδείσους. Ευχαριστώ πολύ την παρακαθήμενή μου αλλά και πολλούς άλλους από άλλες πολιτικές ομάδες που πραγματικά επέδειξαν ε, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και νομίζω ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας ε, μια επιτροπή η οποία εργάστηκε πάρα πολύ συγκεκριμένα, ε, έλαβε υπόψη όλα τα κινήτρα που ερχόντουσαν από όλες τις πλευρές. Έχουμε λοιπόν καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε στα 550 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Σήμερα έχουμε μπροστά μας άλλη μια ευκαιρία για να πούμε ότι πράγματι είμαστε όλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστούμε τώρα η κυρία Ματιού. Eh Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Σαλβατόρε Γιακολίνο, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά και βλέπουμε ότι στέφεται σήμερα με επιτυχία κατόπιν ε, της πιοφορίας αυτής που βλέπουμε ότι ήταν το αποτέλεσμα 29 ψήφοι υπέρ 8 αποχές, καμία ψήφος κατά, μας εξήγησε ο κ. Σταβάρες γιατί υπήρξαν άλλοι που οποία ψήφισαν αποχή. Μεγάλη επιτυχία, όλοι είμαστε εδώ ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες, απαρτία από όλους, ε, καταπληκτικό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Σαλβατόρε για όλη αυτή τη δουλειά που ήταν απαραίτητη ε, και για την ενδιάμεση έκθεση και για την τελική έκθεση. Πάρα πολλές τροπολογίες για τις δύο εκθέσεις. Ε, ήταν πραγματικά τιτάνιο έργο και σε ευχαριστούμε πολύ Σαλβατόρη γιατί το έφερε σε πέρας ε, στο όνομα των συναδέλφων σου. Πραγματικά ε, σου αξίζουν πολλές ευχαριστίες. Επίσης θέλω να απευθύνω τις ευχαριστίες μου και στη γραμματεία, στους συνεργάτες μας που έκαναν επίσης πάρα πολύ δουλειά και σε όλους τους συναντέλφους Επιτροπής ΚΡΙΜ. Ήταν μια προσωπική τουλάχιστον ε, εμπειρία άκρος ενδιαφέρουσα. Για μένα εργαστήκαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτή τη θεματολογία και ελπίζω η τελική έκθεση άποψη και στην Ολομέλεια να αποτελέσει την απαρχή και όχι ε, το πέρας των εργασιών μας. Να είναι μια απαρχή, μια αφετηρία, γιατί θα ψηφίσουμε στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου και ελπίζω σε οποιαδήποτε περίπτωση να αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε και από τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ξέρουμε ότι το έχει ήδη αντιληφθεί η Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα είναι μία μάστιγα. Το ίδιο και η διαφθορά σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αλλά ας μην κρυβόμαστε και σε τρίτες χώρες, αλλά ακόμη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί θα πρέπει σίγουρα να δούμε και τα του οίκου μας. Ελπίζω λοιπόν, Σαλβατόρε, η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα και που αποτελεί καρπό των εργασιών της Επιτροπής μας να ανοίξει το δρόμο και για τους συναδέλφους μας στην προσεχή θητεία. Μακάρι να γυρίσουμε κι εμείς, αλλά αν δεν, επανεξε... Ε, δεν τουλάχιστον η δουλειά αυτή θα έχει γίνει και ελπίζουμε να χρησιμεύσει ώστε να υπάρξει συνδυτοποίηση αλλά και ανάληψη δράσης ε, για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας ε, και γενικότερα της μαφίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και κύριο Σφαγιόν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Σαλβατόρ Γιακολίνου, για όλη τη δουλειά, για την προσπάθεια που αφιέρωσε στην έκθεση αυτή, για την προθυμία που επέδειξε ε, για συμβιβασμό. Να ευχαριστήσω τους κοιόδες, να ευχαριστήσω τους συντονιστές. Νομίζω ότι πραγματικά είμαστε μια εξαιρετική ομάδα αντιμετωπίσαμε σε όλη αυτή την περίοδο διάφορα προβλήματα. παρόλα αυτά καταφέραμε να συνεργαστούμε πολύ καλά παρά τις ε, διαφορετικές μας απόψεις. Πιστεύω Πιστεύω και εγώ, όπως είπε η κυρία Ματιέ, ότι πρόκειται για την απαρχή ε, εδώ στο Κοινοβούλιο μιας ε, εργασίας που θα συνεχιστεί και στην επόμενη θητεία και σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και τη μετάδοση στο, στην κοινή γνώμη όλοι ήταν, είχαν μια πολύ σημαντική συμβολή στην σύνταξη της έκθεσης με την εμπειρία τους. Νομίζω ότι καταφέραμε παίρνοντας και την εντολή για τη δημιουργία ε, του γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, γιατί δόθηκε αυτή η εντολή, καταφέραμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ ρηξικέλεφα κατά την απόψή μου. Βέβαια τώρα θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, να κληθούν να εγκρίνουν ειδικά μέτρα, διότι σίγουρα η έκθεσή μας αποτελεί ε, μια σειρά από συστάσεις, δεν είναι δεσμευτική. Ελπίζω πάντως να εισακουστεί η φωνή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φαγιόν. Και τώρα Αντιπρόεδρος Ταβάρες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να συγχαρώ τον κύριο Γιακολίνο για το έργο του και που υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να συνεργαστούμε. Κατά κύριο λόγο, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Είναι κρίμα βέβαια που χρειαστήκε να απόσχουμε, αλλά νομίζω στην ψηφοφορία της Ολομέλειας να βρεθεί κάποια ισορροπία και κάποια συμβαστική λύση που να μας επιτρέψει να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Μια τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Ταβάρες. Και τώρα ο κύριος Κυλακάκης. Well, uh, uh, thank you, President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πρώτα τον Σαλβατόρη και όλους τους άλλους συναντέλφους που εργάστηκαν πολύ σκληρά και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να δώσω έμφαση ουσιαστικά στο τέλος αυτής της εντολής μας αντέθηκε στο εξής. Για να λειτουργήσει εύρυθμα η Ευρώπη, το ίδιο και για την εύρυθμη του για ναι, Χρειάζεται μια ένωση που θα είναι κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος. Δεν μπορούμε να πετύχουμε στις προσπάθειές μας να έχουμε μια λειτουργούσα ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και σωστά λειτουργούν τα κράτη-μέλη, εάν δεν έχουμε μια ισοδύναμη προσπάθεια στον τομέα της αντιμετώπισης διαφθοράς και του εγκλήματος. Έχουμε θύλακες άκρας διαφθοράς σε πολλά σημεία, σε μέρη που ίσως δεν το περιμένει κανείς. Και αν δεν αντιδράσουμε, η ένωση μας δεν θα είναι ποτέ πλήρης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Μπορκέτσιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να νόσω τη φωνή μου, στη φωνή των υπολείπων, στους επένους και τα εγκόμια που ακούστηκαν, προς τον εισηγητή τον κύριο Γιακολίνο, Απλώς να υπογραμμίσω δύο σημεία. Δύο στοιχεία που ήθελα η Επιτροπή μας να τα έχει πάντοτε υπόψη. Πρώτον, αυτό που ο καθηγητής Κώστα μας επεσήμανε, ένα σήμα συναγερμού που λέει ότι οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές ροές που αφορούν το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών περνούν από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό νομίζω ότι και στην Ολομέλεια θα πρέπει να είναι κάτι που θα το επενθυμίσουμε και έπειτα. Η Επιτροπή αυτή με την έκθεσή της θεωρώ ότι έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει την παρουσία φορολογικών παραδείσων εντός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρουμε όλοι μας πρέπει να επηρεάσουμε με τη δουλειά μας, την πολιτική μας, το πολιτικό μας έργο αλλά και την τεχνική μας δουλειά αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Νιούτον Ντόν. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην Αμερικανική Γερουσία λένε ότι ε, ό,τι πρέπει να υποθεί έχει ήδη υποθεί, αλλά δεν το έχουν πει όλοι ακόμη. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν όλα όσα έπαιρνε προλύσαντες. Απλά θα πω ότι ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να συνεργάζομαι με όλους. Ε, πολλοί είναι εδώ, οι επαγγελματίε, οι σκληροπυρηνικοί αν θέλετε. Χαίρομαι που συνεργάστηκα με όλους σας. Νομίζω ότι κάποιο θα πρέπει να πει και σε εσά κυρία Πρόεδρε ότι την τελευταία ψηφοφορία τη φέρετε σε πέρας με άψογο τρόπο. Δεν υπήρξε καμία διακοπή και ολοκληρώσαμε μέσα σε μια μισή ώρα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Σας είμαι ευγνώμων και όλοι μας είμαστε γιατί φοβάμαστε ότι θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα η ψηφοφορία. Είναι το τέλος ε, της αρχής αν θέλετε γιατί θέλουμε να έχουμε βέβαια καλή, ε, καλό αποτέλεσμα και στην Ολομέλεια. Θέλουμε να υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη δουλειά Θέλουμε η Κομισιόν να πάρει τη σκητάλη, θέλουμε να ενημερωθεί κοινή γνώμη, αλλά και τα κράτη-μέλη να λάβουν δράση και να συμφωνήσουμε στις προτάσεις μας. Άρα παραμένει να γίνει τεράστια δουλειά, αλλά την αρχή ε, την κάναμε. Ευχαριστούμε, Μπιλ, για τα λόγια σου. Ο Αντιπρόεδρος Ντεγιόμ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ και εγώ για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά βέβαια να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά και τον Σαλβατόρη Γιακολίνο. Σαλβατόρη και εσύ έκανες ε, πάρα πολύ δουλειά και έλαβες υπόψη σου και τις δικές μας ανησυχίες ε, στην τελική σου έκθεση. Να πω και εγώ ότι το ότι απήχα τελικά δεν είχε να κάνει τόσο με την έκθεσή σου, αλλά για ένα προεξάρχον ζήτημα, ε, ότι δεν έχει πιστεί ακόμη η ομάδα μου με τα επιχειρήματα της Κομισιόν για ένα γραφείο για Ευρωπαϊκής Αγγελίας, Ευρωπαίου Αγγελέα. Και θα προετοιμάσω και μια σχετική δήλωση για την Ολομέλη, γιατί ιδίω με τις δράσεις προτεραιότητας Νομίζω ότι η έκθεση αυτή πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει στο μελλοντικό έργο που έχει να γίνει στον τομέα αυτό και φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι ότι η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και η νομοποίηση παράνομων εισόδων εισόδων παράνομων δραστηριότητας θα είναι επίκεντρο και στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ. Πριν περάσω και εγώ στα συμπεράσματά μου, να ευχαριστήσω όλη τη γραμματεία και όλο το προσωπικό της Επιτροπής. Το λέω πραγματικά με μεγάλη ικανοποίηση, διότι ήταν η πρώτη μου τέτοια εμπειρία ω ε, Προέδρου, αλλά ευτυχώ που είχα τη συνδρομή τη γραμματεία, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και ο Φιλίπ έχει τώρα το λόγο, γιατί τον ζήτησε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κρηγορήσω. Ήθελα απλά να πω ότι είχα την τιμή και την ευχαρίστηση να είμαι ε, στο, στην κεφαλή μια ομάδα εννιαμελούς, η οποία σα υποστήριξε, προσέφερε τι υπηρεσίε τη στην Επιτροπή σα. Ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ε, και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλου εμά. Δεν θέλω να κάνω λόγο, απλά να σα πω ποιοι είναι οι νέα συνάδελφοι εκτό από τον υποφαινόμενο. Τέσσερι κυρίε. Πλανσόν, ε, Κλέλια Αμπεριαλή, Καρολάιν Οσουλίβαν. Και η κύριοι. Monsieur euh, euh, Andrea euh, Skrimali, euh, Jens Schröder, Yari Erholm et Einars euh, Pungstins, dont je crois au nom. Με τυχαία σειρά, έτσι. Ε, ήταν, ε, νομίζω, ότι ερμηνεύω όλα τα συναισθήματα, μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά για εμά και τιμή που συνεργαστήκαμε μαζί σα. Grazie Philippe. Ehm, Ευχαριστώ Φιλίπ. Ευχαριστούμε για αυτή τη συνεδρίαση αυτή τη Επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με ειδικά καθήκοντα. Όλοι νομίζω ότι ανέλαβαν πλήρω το ρόλο του στα πλαίσια αυτού του θεσμού και να πω ότι στι πρώτε μα συνεδρίασει πολλοί από εσά, του συναδέλφου, έβλεπαν το θέμα αυτό με κάποια απόσταση, δεν θα το έλεγα, αλλά καχυποψία και κάποιου ενδιασμού. Και είχατε δίκιο. Είσαστε υπεπισμένοι κάποιοι από εσά ότι το ζήτημα που εξετάζαμε, το ζήτημα της μαφίας ήταν κάτι που είχε πολύ συγκεκριμένη γεωγραφική ε, σύνδεση με ένα συγκεκριμένο τόπο και γεωγραφικά και οικονομικά και πολιτιστικά. Όμως αυτούς τους 18 μήνες η συνεργασία σας ήταν ε, εξαιρετική. Εμένα δεν μου φάνηκε μακριτό διάστημα των 18 μηνών. Μου φαίνεται σαν να πέταξε ο χρόνος, σαν να πετούσε. Και Πραγματικά βλέπω ότι συνάδελφοι που αρχικά ήταν επιφυλακτικοί, τελικά αγωνίστηκαν, ήταν οι ίδιοι μαχητικοί για να μπορέσουν να ακουστεί η φωνή της Επιτροπής μας και να αφομοιωθεί η άποψη που εκφράζαμε και από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων μας. Ήταν μεγάλη νίκη, ήταν πραγματικά λόγος για τον οποίο δεχτήκαμε συγχαρητήρια ως προς το έργο της Επιτροπής μας και μπορέσαμε πραγματικά να επιβεβαιώσουμε και να συγκρατήσουμε την ε, παρουσία της Επιτροπής μας ως κάτι απαραίτητο ε, που πραγματικά κατάφερε πολλά να πετύχει. Ε, ανέλαβε το καθήκον να εμβαθύνει σε όλα αυτά τα θέματα που σε άλλε επιτροπέ, κυρίω όμω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, λόγω έλλειψη χρόνου αλλά και για άλλου λόγου, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν. Ε, γι' αυτό λοιπόν επανειλημμένω ε, υποστηρίξαμε, αντιμετωπίσαμε και κατανοήσαμε ποια είναι η δικαιότερη τοποθέτηση. Προσπαθήσαμε να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο, όχι μόνο στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά έχουμε 500 500 ε, εκατομμύρια πολίτες σε 27 κρατη και την 1η Ιουλίου φέτο σε 28 κράτη-μέλη. Επισκεφτήκαμε την Ουάσινγκτον, ε, συζητήσαμε από τα τέλη Απριλίου και Αρχής Μαΐου το έργο μας και είδαμε με πόσο ενδιαφέρον οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ ε, κοίταξαν το έργο μας με πολύ μεγάλη περιέργεια αλλά με μεγάλη διάθεση υποστήριξης. Το ακούσαμε να το λέει και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνη, ο κύριος Κόλγεν, που ε, περίμενε με αγωνία το πόρισμα των εργασιών μας, το αποτέλεσμα, δηλαδή τη σημερινή μέρα. Και μας το είπαν και άλλοι Αμερικανοί ηθήνοντε ότι με μεγάλη χαρά όλα τα μέλη της Επιτροπή μα ε, συνετέλεσαν ε, στη δική τους την ε, προσπάθεια εδώ δεν έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα μπει σε ένα σιρτάρι, ένα κείμενο το οποίο θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όχι, ελπίζουμε ότι στην επόμενη θητεία αυτό το κείμενο θα λάβει συνέχεια. Ότι όσα υπόθηκαν σε αυτήν την αίθουσα θα γίνει αντιληπτό σε ένα καθήκον για τους επόμενους, για τους διαδόχους μας, για να αγωνιστούν, να είναι μαχητικοί και να αντιληφθούν ότι το δια, η διαφθορά, η ανακύκλωση και η προώθηση παράνομων ε, εσόδων, αλλά και κατά καταπολέμηση του εγκληματικού εγκλήματο είναι προτεραιότητε. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την ελευθερία και την ε, ευημερία των, πολιτών, των συμπολιτών μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα, ευχαριστώ τον κύριο Γιακολίνο, ευχαριστώ όλου του σκιώδει, όλου του συναδέλφου, τι πολιτικέ ομάδε, του πολιτικού συμβούλου, τη γραμματεία. Σα ευχαριστώ όλου γιατί το έργο πραγματικά αυτό ήταν ομαδικό. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Δεν μπορώ να πω ότι υπερίσχυσε το συμφέρον κάποια πολιτική ομάδα. Με ιδιαίτερη χαρά ε, σημείωσα ότι κανεί δεν προσπάθησε σε αυτή την αίθουσα να προωθήσει τα συμφέροντα επίσης μιας χώρας εναντί κάποιες άλλες. Όχι. Ε, το έργο αυτής της Επιτροπής ήταν έργο που έγινε με σύμπνοια ε, και ελπίζω ότι όλα τα κρατημέλη θα διδαχτούν από τη μέθοδο που ακολουθήσαμε, τη μέθοδο που εφαρμόσαμε στο έργο της Επιτροπής μας, τη δυνατότητα που επιδείξαμε να διαμεσολαβήσουμε, να βρούμε συμβαστικές λύσεις και όχι αποκλει... και αυτό μάλλον προς όφελος της κοινότητας των πολιτών της Ευρώπης, προς το συλλογικό συμφέρον. Από τον Οκτώβριο του 2011, όταν ψηφίστηκε η πρώτη έκθεση για την ε, για τον κατά του είχαμε μια πρώτη ημερομηνία ορόσημο. Σήμερα είναι μια δεύτερη ημερομηνία ορόσημο. Ε, και αυτό θα επαναληφθεί όταν θα ψηφίσουμε στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Το ενιαίο και τελικό κείμενο σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερος, σας ευχαριστώ θερμά, ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστώ μαζί σας, ήταν μεγάλη χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις, έμαθα τόσα, όχι μόνο από την άποψη του οργανωμένου κλίματος, γιατί ακούσαμε τόσους εμπειρογνώμονες, τόσους ειδικούς, Ειδικέ ευχαριστίες προς την Europol, προς όλους τους οργανισμούς που ήρθαν ω εδώ, που ε, μας είπαν ότι ε, γνώριζαν και καθημερινά, ε, άνθρωποι που καθημερινά βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή της ε, μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Έμαθα πόσο σημαντικό είναι να, να, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και να συνεργαζόμαστε και να μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινέ λύσεις. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στην προσπάθεια όλων σας, χάρη στην ατομική προσπάθεια του καθενός και ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε μαζί σας. Ε, το τελικό αποτέλεσμα θα περάσει στα χέρια, για να μην πω στα δάχτυλα των συναδέλφων μας, ε, στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, θα ψηφίσουν και θα μας πούν εάν εργαστήκαμε καλά ή όχι. Πιστεύω ότι θα δείξουν ε, ε, την ικανοποίησή τους. πάντω και πάλι να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς τον εισηγητή. Πάρα πολλέ ευχέ. Θα τα ξαναπούμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Adesso, se non ci sono altre interventi... Αν λοιπόν δεν επιθυμεί κανένας άλλος το λόγο, σας ε, προσκαλώ όλους ε, στη δεξίωση που γίνεται απ' έξω. Είναι το κοκτέιλ δεξίωση που ολοκληρώνει τις εργασίες ε, της Επιτροπής ΚΡΙΜ.